οι διορισμοί αυτοί θα θεωρηθούν εγκεκριμένοι. Η επόμενη συνεδρίαση είναι στις αύριο, στις 22 Οκτωβρίου 2009, από τις 9 έως τη 1 και από τις 3 έως τις 5. Η ημερήσια διάταξη έχει δημοσιευθεί στο ίντρανετ. Ευχαριστώ. Η συνεδρίαση μας έχει λήξει.